Το λόγο έχει ο εισηγητής, κύριο Στέλιτσκα, για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας στο πρόσφατο παρελθόν δεν είχαμε τόσο πολλές ευκαιρίες να επενέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και αυτό. Και οφείλω να πω ότι ο κλάδος της αεροπορίας ήταν μια επιτυχία και μάλιστα χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταστείτε πριν από 20 χρόνια τις αερομεταφορές και τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες για τους καταναλωτές και τους ταξιδιώτες, όλους εμάς. Να πας ένα Σαββατοκύριακο κάπου στην Ευρώπη με φθηνό κόστος ήταν δύσκολο ακόμα και να το φανταστείς. Τότε η αεροπορία ήταν μόνο για λίγους εκλεκτούς. Και σήμερα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα του εννέου ευρωπαϊκού ουρανού και της απελευθέρωσης που καταφέραμε ε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αυξάνονται οι αερομεταφορές και η κυκλοφορία και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και προκλήσεις και προβλήματα. Θα μπορούσα να φέρω ε, περιβαλλοντικούς στόχους σίγουρα. Κανείς δεν θα αρνηθεί σήμερα ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε, να μειώνουμε ε, τις εκπομπές. Ε, ε, ανταγωνισμός με τρίτες χώρες, ψηφιοποίηση. Πάνω από ένα χρόνο τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει φέρει ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε και αυτές και κάποιες άλλες προκλήσεις. Προτείνει να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις με τους βασικούς εταίρους, να αναθεωρήσουμε τους κανόνες ε, για την ΕΑΣΑ, να δούμε ε, επίσης κάποιους εσωτερικούς κανονισμούς. Ε, όλα αυτά είναι πολύ ωραία και ευπρόσδεκτα και έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε από αυτόν, αλλά ταυτόχρονα περιμένουμε και κάποιες νέες προτάσεις. Ο κλάδος των αερομεταφορών χωρίς καμιά αμφιβολία χρειάζεται βαριές επενδύσεις σε ένα περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα. Για να είμαστε αποτελεσματικοί θα πρέπει να έχουμε ένα σαφές όραμα για τις επενδύσεις που κάνουμε σήμερα και για αύριο και να έχουμε γενικότερα ένα όραμα μέχρι με ορίζοντα πέντε αυτό είναι και ο στόχος της έκθεσης, να βρούμε κάποιες πρακτικές εναλλακτικέ προτάσεις για αυτά που σήμερα δεν λειτουργούν σωστά έτσι ώστε να κάνουμε κάποιες ε, προτάσεις για το μέλλον. Δυστυχώς φοβούμαι ότι δεν μπορώ να τις απαριθμίσω όλες, μερικά σημεία μόνο. Πρώτον, ένα δίκτυ διασύνδεσης που να βασίζεται στην προστιθέμενη αξία όλων των τρόπων μεταφοράς, ένα δίκτυ συνδεσιμότητα, όπως λέγεται ε, και να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα και η διασύνδεση παντού στην Ευρώπη. Αυτός ο δείκτης μπορεί να βοηθήσει εκείνου που παίρνουν τις αποφάσεις να πάρουν σωστές αποφάσεις. Ε, δεύτερον, ε, να έχουμε ε, παντού στην Ευρώπη εναέριες λεωφόρους με μείωση των προβλημάτων και να μπορούν απρόσκοπτα οι εταιρείε να κυκλοφορούν. Το έχω συζητήσει αυτό με τους συναδέλφους και υποσχέθηκα ότι θα ξεκαθαρίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ότι στον Ευρωπαϊκό Εναέριο Χώρο θα βάλουμε μια σφραγίδα Ευρωπαϊκή Ένωση όπου θα πρέπει να προηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις πτήσεις της απέναντι στις εθνικές εσωτερικές πτήσεις. Αυτό δεν είναι επέμβαση στην κυριαρχία ούτε τίποτα. Απλώς θυμίζουμε κάποιες υποχρεώσεις που έχουμε κανονικά. Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο αεροπορίας, θα είμαι πολύ σύντομα, να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι θα λύσουμε τα προβλήματα ανταγωνισμού με τις ε, άλλες εταιρείε, ε, βλάπτοντας τον ανταγωνισμό ή σταματώντας τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι και εις βάρος των επιβατών. Βεβαίως να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, αλλά χρειάζεται ανταγωνισμός. Γι' αυτό το Κοινοβούλιο ε, θα παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες. λειτουργικές μεταφορές. Ε, πολύ συχνά όταν μιλάμε για κάποια μέσα μεταφοράς, ιδιαίτερα τα αεροπλάνα, τα βλέπουμε ξεχωριστά από άλλα μέσα μεταφοράς. Και τέλος, ασφάλεια. Δεν χρειάζεται να θυμίσω για ποιο λόγο μας ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό τον καιρό. Βεβαίως χρειάζεται καλύτερος ε, συνδυασμός και συντονισμός των υπηρεσιών πληροφοριών, αυτός ε, υλικοτεχνικός εξοπλισμός ελέγχου και ασφαλείας χωρίς να επιβαρύνονται οι ε, επιβάτες ε, αλλά ένα εθελοντικό σύστημα που να γράφονται εθελοντικά οι επιβάτες έτσι ώστε να περνούν από ένα ειδικό σύστημα ελέγχου στα αεροδρόμια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων το λόγο έχει ο κύριος Κρίστενσεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέρφους της Επιτροπής ε, Μεταφορών και της Επιτροπής Απασχόλησης ε, που προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση στην ε, αεροπορία. Οι κανόνες που έχουμε σήμερα δεν λειτουργούν αρκετά καλά. Κάτι το οποίο είναι κρίμα για τους επιβάτες που είναι θύματα πολλές φορές της συμπεριφοράς αεροπορικών εταιριών. Πρέπει να πούμε ότι οι συνθήκες είναι κακές και ότι γίνεται κατάχρηση κάποιων κανόνων. Πρέπει να διασφαλίσουμε καλύτερη προστασία. Επίσης όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν την κοινωνική τους ασφάλιση, που πληρώνουν φόρους. Χρειάζεται λίγη φαντασία για να βελτιώσουμε την κατάσταση όσον αφορά τους εργαζόμενους στον κλάδο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φροντίσει να υπάρχει συνοχή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κατάλληλε προτάσει για να υπάρχουν ισότιμε συνθήκε εργασία για όλου πρέπει να δράσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, Αλλιώ θα είναι πολύ αργά. Εξ ονόματο τη Επιτροπή, το λόγο έχει η Επίτροπο κυρία Μπούλτ. Good morning. Καλημέρα, καλημέρα Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Σα ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να ανταλλάξουμε απόψει όσον αφορά θέματα αεροπορία και σας ευχαριστώ για την έκθεση πρωτοβουλία σας, η οποία παρουσιάζει μια πλήρη κατάσταση όσον αφορά τον τομέα της αεροπορίας. Ευχαριστώ τον κύριο Τάλισκα, τον κύριο Χρίστιανσεν για την δουλειά τους, όπως επίσης και όλες τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Η αεροπορία φυσικά και έχει σημασία για τους πολίτες μας. Μιλάμε πάνω από 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης άμεσα και πάνω από 100 τόσες θέσεις έμεσα που έχουν να κάνουν σχέση με την αεροπορία. Είναι 6% της παγκόσμιας αγοράς. Γι' αυτό, 26%. Γι' αυτό και χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Είναι σαφές ότι πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έρθω λοιπόν στα βασικά σημεία που αναφέρονται στην έκθεσή σας. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την εσωτερική αγορά. Συμφωνώ απόλυτα την πρόοδο που γίνεται με τους διαφορούς ε, φακέλους που εξετάζεται γι' αυτό. 7 δισεκατομμύρια χάνουμε κάθε χρόνο γιατί δεν προοδεύουμε όσον αφορά τους ενιαίους ευρωπαϊκούς ουρανούς. Επίσης, συμφωνώ με την προσπάθειά σας για την ολοκλήρωση της ενιαία αγορά στον τομέα τη οροπορίας. Επ' αυτού λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτο θα ξεκινήσει μια μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ακριβώς αυτού του ενιαίου ανώτερου χώρου στου ουρανού για να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα των εθέρων μα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση συνεχίζει να στηρίζει τις συμφωνίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αεροπορία και θα σας ενημερώνουμε σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων που κάνουμε. Όσον αφορά τώρα τον ανταγωνισμό του ευρωπαϊκού τομέα αεροπορία, σημειώνω ότι υπογραμμίζεται πω χρειάζονται νέε επενδύσει. Αυτό έχει άμεση σχέση με την συμβασία που έχει ο θεμητό ανταγωνισμό. Εργαζόμαστε λοιπόν σε νέα μέτρα για να προωθήσουμε, να προστατεύσουμε την περιφερειακή ε, συνδεσιμότητα με νέες στρατηγικέ. Περιμένουμε τα νέα μέτρα την άνοιξη και θα συμπεριλαμβάνουν τα εξή. Πρώτον, νέε κατευθυντήρε γραμμέ, όσον αφορά τους κανόνες ε, ιδιοκτησίας για παράδειγμα και μέτρα για την εφαρμογή τους. Δεύτερο, κατευθυντήριε γραμμές όσον αφορά τις υποχρεώσεις των υπηρεσιών. Τρίτον, αντικατάσταση του κανονισμού 868 του 2004 για θέμητες πρακτικές και να τα αντιμετωπίσουμε αυτά με πιο αποτελεσματικά μέτρα. Σκοπεύουμε επίσης να έχουμε και ένα αξιόπιστο μέσο που θα μας επιτρέψει να δρούμε αποτελεσματικά κάθε φορά που οι αερομεταφορεί πλήττονται από πρακτικέ διάκριση ή από θέματα ανταγωνισμού από τρίτε χώρε. Και τέλο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, καταθετήριε γραμμέ για τι ε, υπηρεσίε στον τομέα αυτό. Για τι προδιαγραφέ τώρα. Θέλω να σα πω μερικά πράγματα όσον αφορά την ασφάλεια. Να ξέρετε ότι υπάρχει στήριξη για τον ε, κλάδο αυτό, ιδιαίτερα η ΆΣΑ θα πρέπει να έχει επαρκείς πόρους και επαρκές προσωπικό για να φροντίσει για την ασφάλεια αεροπορίας. Παρακολουθούμε λοιπόν το φάκελο αυτό, ήδη από αυτή τη Δευτέρα έχουμε αρχίσει και ελπίζω ότι θα υπάρξει και νέα ημερομηνία χωρίς νέες καθυστερήσεις. Έχει επιτευχθεί πολύ πρόοδος μέχρι τώρα και είμαι σίγουρη ότι θα ολοκληρώσουμε μέσα στην Μαλτέζικη Προεδρία. Τώρα για το περιβάλλον μετά τη συμφωνία με τον ΙΚΑΟ, τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Είμαστε πολύ σοβαροί στο ότι θέλουμε να πετύχουμε μια αεροπορία με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και θα δώσουμε και οικονομική αρρωγή για να πετύχει αυτό παγκοσμίω. Η αεροπορία είναι μια δραστηριότητα που αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Κανένα δεν μπορεί να μείνει πίσω. Στην ε, πρόταση αυτού του μήνα η Επιτροπή που υφετήθηκε μάλιστα αυτό το μήνα σκοπεύει να φροντίσει για τα συστήματα εμπορίας εκπομπών στην αεροπορία σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Έτσι ώστε να υπάρχουν ισότιμες συνθήκες και ίση μεταχείριση για όλους τους αερομεταφορείς στην Ευρώπη. Για τα κοινωνικά τώρα. Κοινωνική πολιτική ένα τμήμα της έκθεσής σας. Όπως λέμε στη στρατηγική μας για την αεροπορία, Υπάρχουν περίπλοκα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιδιαίτερα έντονη κινητικότητα. Έχουμε δημοσιεύσει τον Μάιο του 2016 κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσουμε τους ε, πιλότους και το προσωπικό ώστε να καθοριστεί το νομικό καθεστώς για τους εργαζόμενους αυτούς που μετακινούνται τόσο πολύ και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει η κατάλληλη ερμηνεία φέτο, ιδίω όσον αφορά την βάση του πληρώματο. Αξιολογούμε λοιπόν το κατά πόσο αυτό, αυτή η έννοια της κύριας κατοικίας μπορεί να εξυπηρετήσει. Συνεχίζουμε την αξιολόγηση του κανονισμού για τα θέματα αυτά και προβλέπουμε να προχωρήσουμε ε, φέτος πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ενισχύσει επίσης τον κοινωνικό διάλογο στην αεροπορία. Ο, η Επιτροπή που ασχολείται με τον κοινωνικό διάλογο πιστεύει ότι θα υπάρξουν νέε ευκαιρίε για του εταίρου μα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να εξολογήσουμε καλύτερα τι κοινωνικέ προκλήσει στον τομέα τη αεροπορία. Ασφάλεια τώρα. Θέλω να είμαι ασφαλή εδώ. Οι ίδιε προδιαγραφέ ισχύουν για όλου, ανεξάρτητα από τι σχέσει απασχόληση. Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα και η ΑΣΕ, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια Αεροπορία, φροντίζει γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να ελέγχουμε τις εξελίξεις στην αγορά και να αναλάβουμε δράση όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Κοινωνικό διάλογο. Αυτό είναι ζωτική σημασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιείται και συνεργάζεται με του κοινωνικού εταίρου, τι χώρε μέλη και όλου του ενδιαφερόμενου για αυτά τα ζητήματα. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Επιτροπή Περιβάλλοντο Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριο Τσάνη. <clears throat> Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θεωρώ πάρα πολύ θετικό ότι οι προκλήσεις των αερομεταφορών αντιμετωπίζονται και όσον αφορά τα δικαιώματα επιβατών αλλά και εργαζομένων. Όλα αυτά τονίζονται στο έγγραφο, αλλά μας τα ε, τόνισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, στην Επιτροπή ΕΝΒΗ θεωρούμε ότι οι αερομεταφορές μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος και να υπάρξουν λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις. Θα πρέπει να αναπτύξουμε με έρευνα και τεχνολογία τις νέες τεχνολογίες προς αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ όλους όσους μας βοήθησαν για την έκθεση της ΕΝΒΗ και τέλος θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα κράτη-μέλη. Ε, να τα ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη, να κάνουν ε, περισσότερα βήματα εφαρμογής ε, των ευρωπαϊκών ουρανών και επίσης να προστατεύσουν τους επιβάτες με σχετική νομοθεσία. και Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε στην Επιτροπή ΙΜΚΟ πέρασε ένα ψήφισμα για καλύτερη προστασία των επιβατών. Σήμερα πολύ συχνά είναι σε αβεβαιότητα οι επιβάτες όταν υπάρχουν προβλήματα με την ε, πτήση τους. Ε, μπορούν να υποβάλουν μια καταγγελία, ε, πώς θα ενημερώνονται, όλα αυτά δεν τα γνωρίζουν πολύ καλά. Επίσης, Όλοι όσοι αγοράζουν μια πτήση επιγραμμικά ή μη θα πρέπει να έχουν την ίδια προστασία γιατί έχουν τα ίδια δικαιώματα και χωρίς να υπάρχουν εξαπατήσεις για τις τιμές των εισιτηρίων. Θα πρέπει να ποντάρουμε σε νέες τεχνολογίες ελέγχου και ε, να έχουμε πρόστιμα αναλογικά ε, με ε, την παράβαση όταν κάποιος δεν τηρεί τους κανόνες. Ως συντάκτρια γνωμοδότηση της ΣΥΜΚΟ λυπάμαι και έχω απογοητευτεί που δεν έχουν ε, συμπεριληφθεί κάποια στοιχεία από τη δική μας γνωμοδότηση για μια στρατηγική μελλοντική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περνούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το λόγο έχει η κυρία Κλούν για 1,5 λεπτό. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Τελίτσια από πλευρά των μελών του ΕΛΚ στην Επιτροπή Μεταφορών για την συνεργασία μας στην ετοιμασία του κειμένου. Τα τελευταία 20-30 χρόνια κάνουμε μια αναδρομή θα δούμε το πόσο ωφέλησε η απορρίθμιση τη αερομεταφορέ. Αυτό είναι σημαντικό για επιχειρήσει, απασχόληση, τουρισμό, συνδέθηκε ο κόσμο, οι περιφέρειε, οι πόλει. Αυτό ήταν τολμηρό, ήταν και φιλόδοξο. Έχουμε και τι εταιρείε ε, χαμηλού κόστου. Τώρα θα πρέπει να πάμε στην επόμενη φάση και έχουμε αυτές τις κατεπίγουσες συμφωνίες για τις αερομεταφορές. Όλα αυτά διατυπώνονται ξεκάθαρα στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σημαντικές οι αερομεταφορές. Ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται τώρα ως προς ειρηνικό, Μέση Ανατολή, τον υπόλοιπο κόσμο. Θα πρέπει επομένως να ε, διευκολυνθούν οι αερομεταφορές γιατί αυτές οι αγορές εξελίσσονται, αναπτύσσονται ταχύως. Είδαμε προς Μαρόκο, προς ε, Βαλκάνια, Καναδά, είπα, έχουν παπλασιαστεί ε, οι πτήσεις και οι δουλειές έχουν ε, αυξηθεί, άρα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε βέβαια το ότι υπάρχει μια περισσότερη κίνηση, αυτό είναι πρόβλημα. Θα έχουμε δύο εκατομμύρια πτήσεις που θα χαθούν γιατί ακριβώς υπάρχει πρόβλημα στα αεροδρόμια. αυτό σημαίνει χρήμα, σημαίνει θέσεις απασχόλησης που θα χαθούν. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους φαγγέλους που είναι ακόμα σε εμπλοκή. Θα πρέπει να υπάρξει επίσης ανθιώρηση του κανονισμού και τα δικαιώματα των ε, καταναλωτών. Οπότε τα πάμε καλά, μπορούμε να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά, αν ενεργήσουμε ταχύως για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις. Για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτον, συγχαρητήρια τον κύριο Ταλίσκα, τον εισηγητή μας, για την υπομονή που είχε προκειμένου διαπραγματευτεί μία έκθεση η οποία προβλέπει το μέλλον πολύ συγκεκριμένα όμως όσον αφορά τον ανώτερο ανέριο χώρο από τη Από την άλλη όμως χρειαζόμαστε, όπως πολύ σωστά είπε, να κοιτάξουμε και τι έχουμε κάνει στο παρελθόν και να δούμε συνολικά την κατάσταση σε μια στιγμή κλειδί που βρισκόμαστε με τόσες αλλαγές στον τομέα της αεροπορίας. Οπότε, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η εκθετική αύξηση των ταξιδιών εξαιτίας του εκδημοκρατισμού στα ταξίδια που έχουμε διαπιστώσει τελευταία οδηγεί και σε κάποια προβλήματα. Σε προβλήματα ικανότητας των αεροδρομίων. Οπότε είναι πάρα πολύ καλέ πολλέ από τις προτάσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται προκειμένου να βελτιώσουμε την ικανότητα αυτή και έτσι να βελτιώσουμε και την συνοχή και τις δυνατότητες των περιφερειακών αεροδρομίων. Άρα λοιπόν προς το μέλλον πρέπει να πάμε σε ομάδες συνδέσεων όπως έχουμε κάνει και με τους σιδηροδρόμους. Είναι ένας τρόπος για να βελτιώσουμε την ικανότητά μας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό και ευχαριστώ που αναφέρεται το κοινωνικό ζήτημα. Και εδώ πρέπει να υπάρξει ισορροπία γιατί η επιτυχία για τους ε, επιβάτες σημαίνει ισορροπία, σημαίνει καλύτερες ηθίκες για τους εργαζόμενους, γιατί θα πρέπει και οι καταναλωτές να έχουν χρήματα για να μπορέσουν να ταξιδέψουν. Άρα λοιπόν μην ξεχνάμε τις επιχειρήσεις και τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις των διαφόρων επιχειρήσεων. Όσον αφορά την τεχνολογία, εδώ χρειαζόμαστε καλύτερη χρηματοδότηση. Στο νέο σύστημα λοιπόν πρέπει, στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να φροντίσουμε να βελτιώσουμε τη χρηματοδότηση και μέσα από το ΕΤΣΕ. Ευχαριστώ πολύ επίσης κύριε Επίτροπε για τον αγώνα που δίνετε εσείς στον ΙΚΑΟ στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να έχουμε κοινωνικά, περιβαλλοντικά πρότυπα και τεχνικά στην Ευρώπη και να τα επιβάλλουμε στον υπόλοιπο κόσμο. Τέλος, πρέπει να υπογραμμίσουμε μια ιδέα που την φέρνω εδώ στο τραπέζι, να υπάρξει ρύθμιση για ανακύκλωση των αεροσκαφών στα πλαίσια της νέας κυκλικής οικονομίας που φέρνει σαν ιδέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Φώστερ. Ε, well, thank you. Thank you. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κυρία Επίτροπε. Πρώτα πρώτα θα πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμότατα τον Παύλ Τελίτσκα γιατί ήταν εξαιρετική η εργασία που έκανε όσον αφορά την έκθεση για τις αερομεταφορές 99% επομένως παίρνει άριστα και θα τον υποστηρίξουμε. Όμως προέκυψε κάποιο σοβαρό πρόβλημα γιατί η Επιτροπή Απασχόληση είχε αποκλειστική αρμοδιότητα ε, σύμφωνα με το άρθρο 54 όσον αφορά τα γεωνικά θέματα. Αλλά όσον αφορά εδώ τους πιλότους των αερομεταφορών συμβαίνει το ότι έχουν κάποιες συμβάσεις παράνομες. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τους επιβάτες. Ε, αυτό καταγνωρίζουν τα στοιχεία. Και έχουμε επίση για το επιχειρηματικό μοντέλο όσον αφορά επίσης την έδρα των εταιριών, κάποια προβλήματα και άρα εδώ αγνοούνται αυτά τα φαινόμενα. 70% των πτώσεων των, πτήσεων στην Ευρώπη αφορούν αυτές τις αερομεταφορές και έχουμε τις, τα πιο αυστηρά στάνταρ όσον αφορά τις συμβάσεις, όσον αφορά τους πιλότους, τα πληρώματα, ε, τους περιορισμούς για τον χρόνο πτήσης, οπότε υπάρχουν κατηγορίες οι οποίες όμως είναι αστήρικτες και ακόμα χειρότερα δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό το οποίο έπρεπε με την Επιτροπή Απασχόληση. Θα πρέπει να υπάρχουν καλέ συνθήκε απασχόληση, θα πρέπει να υπάρχει κατάρτιση, αλλά όλα αυτά δεν περάσαν στην έκθεση. Εμεί θέλουμε όλα αυτά, σωστέ συμβάσει, δίκαιε δηλαδή. Και επομένω τώρα θα στείλουμε το λάθο μήνυμα. Θα κακό για την Επιτροπή Απασχόληση. Αυτή θα πούμε ότι δεν πρέπει οι Ευρωπαίοι να πετούν ευρωπαϊκές εταιρείες. Μα είναι ντροπή. Οπότε εγώ δεν μπορώ να συνενέσω με τέτοια πράγματα που λέει η έκθεση και δεν μπορέσαμε να τα αλλάξουμε. Και πάλι βέβαια, ε, μπράβο στον κύριο Τέλτσκα, νομίζω με καταλαβαίνει και ελπίζω το καταλάβατε αυτό που λέει ο κυρία Επίτροπε. Να προσέχουμε πάρα πολύ όταν επιτρέπουμε σε άλλες επιτροπές να συμβάλλουν τόσο πολύ για κάποια ζητήματα. Προσοχή, δεν είναι σωστό αυτό. Θα έπρεπε μια γνωμοδότηση να αρκεί. Το λέει αυτό η Επιτροπή Μεταφορών, γιατί είναι θέμα μεταφορών. Και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ομάδα των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει πολύ καλή πρόταση για τη στρατηγική στην Ευρώπη και τώρα έχουμε μια πολύ καλή έκθεση για τη στρατηγική του Παύλ Τέλιτσκα και θέλω να τον συγχαρώ. Ε, ο πληθυσμό τη γη αυξάνεται και γεμίζει όλο και περισσότερο ο εθέρα, όχι μόνο γιατί μεταφέρονται ε, αλλά και ε, προϊόντα. Ε, Μιλάμε για λεωφόρους. Ε, λεωφόρους έχουμε ε, αυτοκινητοδρόμους, έχουμε πλέον θαλάσσιες και αέριες, παρόλο που δεν κυκλοφορούν αυτοκινήτα, αλλά αεροπλάνα και χρειάζεται χώρος για να ε, κυκλοφορούν διάφοροι. Και δεν πρόκειται μόνο για μεγάλα αεροσκάφη επιβατηγά, έχουμε και μικρά ιδιωτικά jet drones και πάει λέγοντας. Χρειάζεται ένας ανταγωνισμός υγιής και θεμητός, όχι μόνο μεταξύ των ε, διεθνών αερολιμένων. Η Φραγκφούρτη έχει τη σημασία της, ε, αλλά την έχει χάσει ως κόμβος, την έχει ξεπεράσει η Κωνσταντινούπολη. Στις αεροπορικές εταιρείες υπάρχουν πάρα πολλές ε, ε, πρακτικές ανταγωνισμού. Βεβαίως χρειάζεται καινοτομία, θα πρέπει να είμαστε πιο φιλικοί προς το ε, περιβάλλον. Ε, περιμένω το πρώτο αεροσκάφος το οποίο θα καταναλώνει τα καύσιμα που θα παράγει μόνο του στην κυκλική οικονομία και τέλος χρειάζονται και σωστοί κανόνες για τα κοινωνικά, για τα εργασιακά, για τα δικαιώματα των επιβατών και ένα ευρωπαϊκός ε, ουρανός χρειάζεται και συνειδητά τελειώνω με αυτό. Έχει μπλοκαριστεί ε, εδώ και δύο χρόνια αυτό το θέμα. Πετάμε ζυγζάκα αντί να έχουμε συνδέσεις ευθεία στον ουρανό μας. Τι θα γίνει, επιτέλους θα έρθει αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Κονέτσνα. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πολύ για την έκθεση αυτή. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον εισηγητή από την αρχή. Είχε κάποιες θέσεις, αλλά έκανε και υποχωρήσεις και έλαβε υπόψη τα κοινωνικά ζητήματα στην έκθεσή του. Αυτό έγινε μετά από πίεση της Επιτροπής Απασχόλησης, αλλά και από πιέσεις άλλων συναδέλφων θέλουμε να λαμβάνονται υπόψη και οι υπηρεσίε και τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που λέγει η συνάδελφο Φώστερ. Καλό είναι να γνωμοδοτούν και άλλε επιτροπές. Με ιδιαίτερη χαρά βλέπω ότι η έκθεση αναφέρεται στην ΕΑΣΑ και στα κράτη-μέλη και καλούν καλούμε στην έκθεση να βρούμε νέα μοντέλα επιχειρηματικά πτήσης και απασχόλησης των εργαζομένων. Ιδιαίτερα τη συμβάσει μηδενικών ωρών πρέπει να κοιτάξουμε γιατί είναι άδικες απέναντι στους εργαζομένους. Εγώ είμαι υπέρ μιας ισχυρής ευρωπαϊκής αεροπλοείας αλλά δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος των εργαζομένων σε αυτήν. Θα πρέπει αυτά τα θέματα να τα συνδέσουμε, να τα γνωρίζουμε και το καταφέραμε στην έκθεση. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ. Για την ομάδα των Πρασίνων το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Νταλούντε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η κυκλοφορία με τις αερομεταφορές όλο ένα και αυξάνεται τη σημερινή μέρα και αυτό είναι κάτι το θετικό γιατί έχουν περισσότερη κινητικότητα, όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι εκπομπές από τις αερομεταφορές επίσης ε, αυξάνονται και αυξάνεται η βλάβη προς το περιβάλλον. Επίσης θα πρέπει να συγκρατήσουμε αυτές τις εκπομπές για μας τους πράσινους είναι πάρα πολύ σημαντικό οι αερομεταφορές όπως και οι υπόλοιπε μεταφορές να πληρώσουν για τις συνέπειες που υπάρχουν εις βάρος του περιβάλλοντος. Έχουμε το ETS, ε, έχουμε τεχνολογίες, ε, έχουμε διάφορους τρόπους ε, επένδυσης, έχουμε κάποιες πράσινες προσεγγίσεις, αλλά δεν αρκούν αυτά. Χρειάζονται κάποιοι κανόνες για να είναι έχουμε κάποιες ανταγωνιστικές εναλλακτικές. να έχουμε ας πούμε τρένα ψηλής ταχύτητας, να έχουμε διαφορά δίκτυα, νυχτερινά τρένα, βιώσιμα καύσιμα για τις αερομεταφορές. Είναι παράδεκτο για αερομεταφορές να μην πληρώνουν για τις ε, συνέπειες της δραστηριότητάς τους. Έχουμε ένα σωρό αεροδρόμια τα οποία επιδοτούνται με τα χρήματα των φορολογουμένων. Αυτά δεν είναι σωστά. Χθε ψηφίσαμε για την μεταρρύθμιση του ETS, του Συστήματος Εμπορίας των Εκπομπών και θα πρέπει να σκεφτούμε τι γίνεται και με τις αερομεταφορές, τι γίνεται με το περιβάλλον. Τελικά η μεταρρύθμιση αυτή ήταν απονευρωμένη. Έτσι δεν πρόκειται να πετύχουμε αυτό που συμφωνήσαμε στο Παρίσι. Άρα θα πρέπει το κόστος της βάρος του περιβάλλοντος να αντισταθμιστεί από τις αερομεταφορές. Να μην κοιτούμε το κοντόφθαλμο όφελος. Την ομάδα Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας. Το λόγο έχει για δυόμιση λεπτά ο κύριος Πάξας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση αποτελεί μια θετική εξέλιξη και από ό,τι γνωρίζω η στρατηγική, η πολιτική για τις αερομεταφορές αφορά ανταγωνιστικότητα, αφορά ασφάλεια, αφορά και τα θέματα των ενιαίων ευρωπαϊκών ουρανών και από ό,τι γνωρίζω έχουμε τις προτάσεις Τέλιτσκα οι οποίες ε, αποσκοπούν στο να υπάρχει περισσότερη ασφάλεια επίσης κάτι το οποίο χρειάζεται και η ευρωπαϊκή πολιτική για τις αερομεταφορές θα πρέπει να οδηγήσει ανταγωνιστικότητα, να δούμε τι θα γίνει, να μπορέσουμε να έχουμε στη διεθνή σκηνή κάποια κυριαρχία, κάποια δεσπόζουσα θέση. Τα μικρά αεροδρόμια θα πρέπει να τα προσέξουμε να γίνουν προτεραιότητα. Νομίζω ότι αυτό το ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχουν κάποια οικονομικά μέτρα από τα κράτη-μέλη ώστε να επιβιώσουν αυτά τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια κυρίως στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πάνω από 40 χρόνια έχω δίπλωμα πιλότου και παρόλα αυτά κύριε Τελίτσκα έχω κάποια προβλήματα με το κείμενο όπως και άλλοι που ασχολούνται με τις αερομεταφορές. Γιατί ενώ μας απασχολεί η ανεργία των νέων δεν κάνουμε κάτι για τα αεροδρόμια και την πτήση που αφορά και αθλητικές ε, εκδηλώσεις θα πρέπει να υπάρξει έλεγχος, ρύθμιση, είναι θέμα κρατικό, δημόσιο. Τι θα γίνει με τα αεροπλάνα, τα διθέσια, τα τετραθέσια, τα ιδιωτικά. Να υπάρξει ρύθμιση για όλα τα αεροδρόμια και όχι μόνο για τα Boeing οι αεροναυπηγοί κατασκευάζουν ασφαλή αεροπλάνα. Εμείς όμως από την άλλη μεριά χάνουμε το χρόνο μας στους ελέγχους ασφαλείας. Γιατί τόσες καθυστερήσεις. Τελικά δεν είναι πρόβλημα μόνο οι καιρικέ συνθήκες. Θα πρέπει να προστατευτούν οι καταναλωτές. Τι γίνεται επίσης με τη ζημία ει βάρος των κατανοτών από τις απεργίε των αερομεταφορών. Προσοχή, να δούμε πώς θα το αντιμετωπιστούν στο μέλλον. έχει 3,5 λεπτά η κυρία Αρνοτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, πάνω από 30 χρόνια έχω δουλέψει στην Air France και δυστυχώς διαπιστώνω τα προβλήματα από τον υπερβολικό ανταγωνισμό στον τομέα της αεροπορίας. Θέλοντας να κάνουμε υπερβολικά πολλά, να απορριθμίσουμε λόγω του κέρδους, η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά οδήγησε σε ένα πλαίσιο από το οποίο υποφολούνται πολύ περισσότερο οι ξένες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους παρά οι εθνικές παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες δυσκολεύονται είναι σαφές. Είτε πρόκειται για τους μεγάλους παραδοσιακούς αερομεταφορείς, είτε για τα αεροδρόμια. Αυτός ο ανταγωνισμός γίνεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο η αεροπλοεία μπορεί να κερδίσει κάπως. Τι έχουμε να πούμε όμως για την Airbus η οποία μεταφέρει τις δραστηριότητές της, μειώνει τον προπολογισμό της για την έρευνα και την ανάπτυξη και μειώνει και το προσωπικό. Επίσης, Διαφωνώ με αυτό που αναφέρει ο εισηγητής για τον απαράδεκτο ανταγωνισμό. Εγώ νομίζω ότι εδώ είναι η αντίθετη λογική που πρέπει να υπερισχύσει. Όπως και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εδώ και 40 χρόνια που έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται οι ελεύθερες συναλλαγές δόγμα υπέρ μιας, ενός άκρα του ανταγωνισμού ακόμα και στον τομέα της αεροπορίας που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αθέμητο ανταγωνισμό από τις χώρες του κόλπου. Αλλά, κύριε Σιγητά, δεν με εκπλήσει και τόσο πολύ που εσείς συμφωνείτε με αυτήν την μερκατιλίστικη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί και εσείς εκεί ήσασταν ε, πριν. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι θα έπρεπε οι δημόσιες αρχές να υποστηρίζουν την απασχόληση των δικών τους υπηκών και να προστατεύουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Και αν κάποιοι πιστεύουν ότι ο προστατευτισμός στον τομέα της αεροπορίας είναι λαϊκισμός, τότε εντάξει, ευχαρίστω, το παίρνω και σαν κομπλιμέντο. Δεν θα έπρεπε να εξαφανίζονται τόσες επιχειρήσεις ή να συγχωνεύονται με άλλες διεθνεί επειδή το κράτος δεν έχει το δικαίωμα να τη σώσει, ούτε θέλω τη συγχώνευση αυτού του καινούριου business ε, model που καταλήγουμε σε αεροπορικές εταιρείε, απλώς και μόνο θηρίδα και τίποτα άλλο. Οι συστάσεις της Επιτροπής ε, Απασχόλησης με ικανοποιούν αλλά περιμένω την βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τις εφαρμόσει όλα και όχι να τιμωρεί τέτοιες συμπεριφορές παρόλο που έχουν να κάνουν με την προστασία την ίδια των επιβατών. Καμία χαμηλού κόστος αεροπορική εταιρεία δεν είναι στις 10 πρώτες αεροπορικές εταιρείες ε, κατάταξης. Άκουσα τον εισηγητή, δεν με πείθει. Θα κρατήσω θέση αποχής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό, ο κύριος Ζαριανόπουλος, μία εγγεγραμμένος. τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό τη στρατηγική αερομεταφορών της ευρωπαϊκής ένωσης για ιδιωτικοποίηση υποδομών υπηρεσιών και του εναέριου χώρου βιώνουμε και στην ελλάδα με την παράδοση από την κυβέρνηση σύριζα ανέλ σε συνέχεια του προηγούμενων δεκατεσσάρων αεροδρομίων στην κοινοπραξία φραπόρτ κοπελούζου. οι εργαζόμενοι τη πολιτική αεροπορία όλοι οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια μένουν κυριολεκτικά στον αέρα μη γνωρίζοντα αν θα έχουν δουλειά και δικαιώματα. η ασφάλεια των πτήσεων με τη λογική κόστου ωφέλου τίθεται σε κίνδυνο. ο τουρισμό που εξυπηρετείται από τα αεροδρόμια παραδίδεται σε συνδεδεμένου μεταφορικού και τουριστικού ομίλου κρατικές υπηρεσίες όπως η πυροσβεστική τίθενται στην υπηρεσία του ιδιώτη. παραδίνεται ο έλεγχος του εθνικού εναέριου χώρου σε ιδιωτικά μονοπόλια πολλαπλασιάζοντας τους κινδύνους για ζωτικά κυριαρχικά δικαιώματα της ελλάδας σε μια περιοχή το αιγαίο και σε μια χρονική περίοδο που αυτά αμφισβητούνται ευθέως από την τουρκική ηγεσία με καθημερινή αμφισβήτηση των συνόρων εναέριων και θαλάσσιων και τη συνθήκη τη λοζάνη που τα καθορίζει. ο λαό να σταματήσει την παράδοση των αεροδρομίων ενιαίος δημόσιος φορέας αερομεταφορών για τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα μονοπωλιακά κέρδη. Επόμενος ομιλητής για 1,5 λεπτό, ο κύριος Βαντεκάμπ. Ε, <clears throat> Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Πρώτον, ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για την έκθεση αυτή. Πιστεύω ότι δίνει μια πολύ καλή εικόνα αυτού που θέλουμε να κάνουμε με την αεροπορία στην Ευρώπη. Και είναι σαφές και υπόθηκε κιόλα ότι πρόκειται για ένα τομέα που αποτελεί μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Είναι ένας τομέας που ελευθερώνεται. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες τώρα μπορούν εύκολα, πιο εύκολα από παλιά να πετάξουν, να πάνε διακοπές. Θέλω να αναφέρω τέσσερα ζητήματα. Πρώτον, την δύναμη καινοτομία του τομέα αυτού. Η Επιτροπή Μεταφορών την επόμενη εβδομάδα θα πάει στην Τουλούζη. Θα επισκεφθεί την ε, Airbus και θα δει εκεί τι γίνεται με αυτή την καινοτομία στην Ευρώπη. Δεύτερον, Πρόεδρε, ανταγωνισμός. Πράγματι, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός ε, βαρύ στον τομέα. Δεν είναι πάντα εύκολο και απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτο θέμα, κοινωνικά ζητήματα παρακολουθούμε το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να μην λαμβάνουμε υπόψη μας την απασχόληση. Και τέταρτον, νέοι πιλότες. Πρέπει να τους προσέξουμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Ντεμόντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κυρία Επίτροπε. Οι αερομεταφορές είναι κλειδί για τις μεταφορές. Θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση έτσι για τις συνδέσεις μέσα και έξω από την κοινότητα. Χρειάζεται επομένω στρατηγικός προγραμματισμός όσον αφορά το σύστημα των αεροδρομίων στην Ευρώπη. Και έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για όλα τα αεροδρόμια και τα περιφερειακά απασχόληση να δημιουργηθεί, να βοηθηθεί ο τουρισμός και επομένως να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την κυκλοφορία στα βασικά αεροδρόμια αλλά να βοηθήσουμε και τις πιο μακρινές περιοχές. Τα λέει αυτά η ανακοίνωση της Επιτροπής για κάποιες ενισχύσεις όσον αφορά τη βοήθεια του κόσμου για τα μικρά αεροδρόμια τα οποία έχουν σημασία ε, τοπική. Και για αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβούμε σε επενδύσεις και έτσι να ε, έχουμε ενισχύσεις, να έχουμε επενδύσεις γιατί θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη αξιοποίηση των αεροδρομίων και από εμπορική πλευρά. Που έχει για 1,5 λεπτό ο Βαντάλεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην αρχή ο κύριος Τέλετσκα έδωσε βάρος στην καινοτομία και στην ε, συνδετικότητα αλλά και στον ανταγωνισμό. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερα τα προβλήματα στις αερομεταφορές. Είναι μια κούρσα για ε, την πιο μικρή τιμή και την πληρώνουν οι κυβερνήτες. Τώρα πρέπει να πληρώνουν για να μπορούν να πετάνε. Pay to fly λέγεται αυτό το σύστημα, είναι γνωστό. Και αυτό είναι πρόβλημα και για τους κυβερνήτες και για τους ε, ε, επιβάτες, αλλά φαίνεται ότι είναι ένα μοντέλο του London School of Economics. Ε, οι πιλότοι διαμαρτύρονται για υπερκόπωση, δεν τους λαμβάνουν υπόψη οι εταιρείε. Αυτό είναι ένα παράλογο σύστημα το pay to fly και δείχνει μια κουλτούρα ε, οργάνωσης με μεγάλα ρίσκα και κινδύνους. Και διάφορες οργανώσεις και συνεργατικές οργανώσεις κυβερνητών έχουν αρχίσει να ε, κινούνται ε, δικαστικά και σωστά απέναντι σε τέτοια συστήματα. Ευτυχώς ο εισηγητής το κατάλαβε και το έβαλε πλέον στην έκθεσή του αυτό, το υιοθέτησε και χαίρομαι. Και με τις αλλαγές και τις προσαρμογές μπορεί τώρα να υπερψηφίσω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Κίλονεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να μας πει η Επίτροπος τι γίνεται με τα βιοκαύσιμα. Ιδίως όσον αφορά την δεύτερη γενιά βιοκαυσίμων χρησιμοποιούνται από τις αερομεταφορές για να έχουμε έτσι μείωση των εκπομπών. Εμείς θέλουμε να υπάρχει χρήση τέτοιων βιοκαυσίμων, όμως πολλές φορές η τιμή τους φτάνει μέχρι και τρεις φορές πιο ακριβή από ό,τι των παραδοσιακών καυσίμων. Άρα, θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι για να πετύχουμε τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται και από τι αερομεταφορέ και από τι καταθάλασσε μεταφορές. Και γι' αυτό ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κατευθυνθεί προς τα εκεί. Να μπορέσουμε να μην εξαρτώμεθα από τα ρηκτά καύσιμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή μας, τον κύριο Ταλίσκα. Η αεροπορία είναι ένας τομέας με μεγάλο δυναμισμό. Όσον αφορά εκπομπές διοξοδίου του άνθρακο, όμως μέχρι το 2050 θα πολλαπλασιαστούν εκπομπές επί 7. Ήδη ο τομέας αυτός είναι 3% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα παγκοσμίω. Οπότε από μόνος του ο τομέας της αεροπορίας θέτει σε κίνδυνο τους στόχους του COP21. Για μένα δεν υπάρχει περιθώριο για τέτοιες εξελίξεις. Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στην τεχνολογία. Και πέρα από το θέμα του κλίματος υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Ότι είναι απορριθμισμένο ο τομέας. Έχουμε έναν αθέμητο ανταγωνισμό με τα τέλη ε, αερολιμένων, με τις αεροπορικές εταιρείες του κόλπου. Πρέπει να κάνουμε όπως και στους σιδηροδρόμους. Η κυροζήνη δεν φορολογείται. Πρέπει επίσης να κοιτάξουμε και την απασχόληση στο τομέα αυτό με το pay to flight, με τις υπερβολικές ώρες απασχόλησης των πιλότων. Πρέπει να δούμε λοιπόν και την ασφάλεια και τα κοινωνικά ζητήματα. Άρα είναι ένας τομέας ο οποίος πρέπει να λάβει υπόψη του το περιβάλλον, το κοινωνικό αλλά και το τεχνολογικό φάσμα. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Προύστ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η αεροπορία και ο ναυπηγικός ε, τομέας, εκατοντάδες ε, χιλιάδες εργαζομένους έχουν σε άμεσες 190.000 στη Γαλλία και είναι πυλώνας ανάπτυξης. Αυτό το είχε καταλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν το Δεκέμβρη του 2015 κατέθεσε ανακοίνωση για μια στρατηγική. Σήμερα συζητούμε το σύνολο της έκθεσης που είναι πλήρης, λαμβάνει υπόψη της όλα τα στοιχεία έτσι ώστε να ενισχυθεί η Ευρώπη και στην εσωτερική αγορά και στη διεθνή. Ασφάλεια στην ενέργεια κυκλοφορία με μεταρρύθμιση άσα, ενιαίος ουρανός, δικαιώματα επιβατών, συμφωνία για τις εκπομπές και διεθνής ε, πτυχή. Όλα αυτά είναι άξονε προτεραιότητας που θα πρέπει να κατευθύνουν και να καθοδηγούν κράτη-μέλη και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πέρα από την ίδια τη στρατηγική όπως και στα αθλήματα αγωνίζομαι να υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες παντού. Δυστυχώς υπάρχουν αθέμητες πρακτικές ακόμα, εμπορικές πρακτικές. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε και τις εταιρείε μας και τους ερωλημένες μας. Γι' αυτό κύριε Επίτροπε να μεταρρυθμίσετε σωστά τον κανονισμό για τις αθέμητες πρακτικές και τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο κλάδος να ε, ξαναβρει προοπτικές γερές για το μέλλον του. Ευχαριστώ το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Άντερσον. Good morning, everyone. Um, the continuing success... Καλημέρα σας. Η... Σημαντικό να συνεχιστεί η επιτυχία μας όσον αφορά τις ευρωμεταφορές και για τους εργαζόμενους και για τους ε, επιβάτες. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δουλεύουν πάρα πολύ ε, καλά όσον αφορά την καινούργια γενική στρατηγική. Θα πρέπει επομένω να δούμε τι θα γίνει, να συνεργαστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα καινούργιο πλαίσιο ρυθμιστικό για αυτόν τον κλάδο. Για να έχουμε ε, ένα κοινό όραμα, ο Ευρωπαϊκό Ουρανό να υλοποιηθεί πέραν των εθνικών αποκλήσεων αυτό ωφελεί όλου και να κάνουμε επομένω ό,τι πρέπει από το χέρι μα, ούτως ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχει σε ε, αυτό το όραμα στο μέλλον. Τώρα για τις ε, λεπτομέρειε όλοι οι βουλευτές θα πρέπει να κάνουμε κάτι ούτω ώστε να μειωθεί, να συγκρατηθεί η ζημία στο περιβάλλον. Θα πρέπει να γίνει μια στροφή προς άλλε μεταφορέ όπου γίνεται αυτό οπότε θα έπρεπε η έκθεση να τα λέει καλύτερα. Αλλά τέλο πάντων εγώ θα, θα την ψηφίσω την έκθεση Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και αντίθετα με το ότι είπαν κάποιοι άλλοι συναδελφοί, περισσότεροι συμφωνούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, ότι υπάρχουν προβλήματα για εργαζόμενους, ε, για το, ε, για το προσωπικό εδάφος και για τους πιλότους. Θα πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Κύριος Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η αεροπορία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τη δημιουργή ανάπτυξη και απασχόληση και καινοτομία στην Ευρώπη. Συνεπώς η στρατηγική μας αυτή δικαιολογείται απόλυτα. Οι αεροπορικές εταιρείες και οι πολωνικές δημιουργούν πλούτο, έσοδα και ανταγωνίζονται καλά στην παγκόσμια αγορά. Χρειάζονται όμως ακόμα συστήματα διευκόλυνσης και διμερών συμφωνιών. Χαίρομαι λοιπόν που ο κύριος Ταλίτσκα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην διαθεσιμότητα αερομεταφορών και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ περιφερειών και χωρών μελών. Όσον αφορά το σημερινό επίπεδο προσβασιμότητας, το να χρησιμοποιούνται φτηνές διασυνδέσεις κοντά στο χώρο κατοικίας κανενός είναι πάρα πολύ θετικό και μπορεί να διασφαλιστεί χάρη στον κατάλληλο ανταγωνισμό στον τομέα των αερομεταφορών και επενδύοντας και στις υποδομές. Το μέλλον της οροπορίας λοιπόν πρέπει να λάβει υπόψη την ασφάλεια των επιβατών ως προτεραιότητα, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό το επιχείρημα να το χρησιμοποιούμε για τα πάντα και για τις ε, τσακωμούς μεταξύ υπαλλήλων και εργοδοτών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πήρα το λόγο για να σας ζητήσω να υπερψηφίσετε την τροπολογία 2 μετά την παράγραφο 15 που αναφέρεται στην ακύρωση της παραχώρησης 14 κερδοφόρων περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα υπέρ της Φράμπορντ. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση απικιακής σύμβασης. Είναι αποτέλεσμα πολιτικού εκβιασμού καθώς ετέθη ως προαπαιτούμενο για την υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Παραβιάζει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμός. Τεχνικός σύμβουλος της διαδικασίας παραχώρησης ήταν η εταιρεία lufthansa που είναι μέτοχος της fraport. η ίδια η fraport κατά μεγάλο ποσοστό ανήκει στο γερμανικό κρατήριο της ΕΣΥ με συνέπεια αυτή η συμφωνία να είναι παραχώρηση δημόσιας περιουσίας ενός κράτους μέλους σε ένα άλλο κράτος μέλος. συνολικά οι όροι της σύμβασης εξαιρούν την εταιρεία από μια σειρά δεσμεύσει και υποχρεώσει οικονομικού ε, οικονομικών υποχρεώσεων στο ελληνικό δημόσιο στους εργαζόμενους και στις τοπικές δημοτικές αρχές. αγαπητοί συνάδελφοι αν θέλουμε να σταθεί στα πόδια του ελληνικό ελληνικός λαός δεν θα το κάνουμε αφαιρώντας τη δημόσια περιουσία. γι' αυτό σας καλώ και πάλι να υπερψηφίσετε αυτή την τροπολογία που ζητάει την ακύρωση αυτής της απικιακού τύπου σύμβασης που έχει δρομολογηθεί. ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θέλω να πω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πάντα ισχυρίζονται ότι έχουν συνολικές προσεγγίσεις για κάθε είδους πρόβλημα. Από τη Γενική Διεύθυνση μου είχαμε εκθέσεις ωραίες, στρατηγικές για το μέλλον των μεταφορών. Άμα πας όμως κλαδικά εκεί θα δεις ότι χάνεται η συνολική προσέγγιση. Η στρατηγική για τις αερομεταφορές είναι πραγματικά μονομερής προσέγγιση. Κοιτάει μόνο τα προβλήματα του αθέμητου ανταγωνισμού διεθνώς και κάποια ζητήματα που έχουμε και στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Δυστυχώς ο εισηγητή Επίση επίσης δεν ε, έχει μια καθολική πραγματική προσέγγιση που χρειάζεται ο κλάδος και χαίρομαι που στον κοινωνικό πυλώνα διορθώθηκε και βελτιώθηκε η έκθεση αυτή. Ωστόσο, ε, στα περιβαλλοντικά σχεδόν τίποτα δεν κάνει. Δεν αναφέρει καν τη Συμφωνία των Παρισίων. Και όταν όλοι διαρριγνύουν τα ημάτια του και πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά, όταν συζητούμε αυτό τον κλάδο δεν αναφέρεται καθόλου. Τι δείχνει αυτό, ότι η καθολική προσέγγιση λείπει και όταν πάμε στα κλαδικά λέμε ότι πρόκειται ε, για οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Εγώ θα καταψηφίσω την έκθεση, δεν με καλύπτει. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Λόπες Μπερμέχο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι αερομεταφορές είναι όπως και άλλοι κλάδοι θύμα των απορριθμίσεων και των ιδιωτικοποίησεων τη Κομισιόν και των κρατών μελών και στην Ισπανία ισχύει αυτό η ΑΕΝΑ έτσι γίνεται η διαχείριση και τελικά το, το κέρδος είναι για τις εταιρείες εις βάρος όμως των εργαζομένων και των επιβατών. Οπότε είχαμε σαφώς επιδίνωση για τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο αυτό. Οι υπηρεσίε αυξήθηκαν κατά 47% τις τελευταίες δεκαετίες, όμως δεν βελτιώνεται η απασχόληση και έχουμε κάποιες προσωρινές συμβάσεις, έχουμε τις μηδενικές συμβάσεις και όλες αυτές είναι ευάλωτες και αυξάνονται. Θα πρέπει να ακούσουμε τι λένε τα συνδικάτα, να γίνουν συλλογικές συμβάσεις και να δούμε τι αλλαγές θα πρέπει να γίνονται όσον αφορά τις συμβάσεις και παραχωρήσεις αεροδρομίων. Δεν θα πρέπει να συνεχιστεί η επιδείνωση των εργασιακών συνδικών, να σταματήσει το κοινωνικό dumping, να σταματήσουν οι ιδιωτικοποίησεις. Ε, ολοκληρώσαμε τη διαδικασία με τους εγγεγραμμένους ομιλητές. Προχωρούμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Έχω δεχθεί πέντε αιτήματα. Θα κάνω και τα πέντε αποδεκτά. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ. Είμαστε ευγνώμονες στις αεροπορικές εταιρείες που μας φέρνουν εδώ κάθε εβδομάδα στις Βρυξέλλες και θέλω να ευχαριστήσω και την Air Lingus για την αποτελεσματικότητα με την οποία εργάζεται. Τώρα οι διαπραγματεύσεις για το Brexit προχωρούν και ένα σκληρό Brexit θα οδηγήσει σε προβλήματα στην αγορά του κλάδου και όχι μόνο. Εξαιτίας λοιπόν μεγάλων δυσκολιών στις ε, μεταφορές υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τις θαλάσσιες μεταφορές, ε, τις εμπορικές. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και συμφωνώ με τον ναδερφού Eichhout και άλλους ότι η συμφωνία των Παρισίων πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε την αύξηση στη ζήτηση, αλλά να μειώσουμε τις εκπομπές. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θέλω να συγχαρώ τους συζητητές και όλους όσοι συνεισέφεραν στην έκθεση αυτή. Ε, Ξέρω τι συμβαίνει στην Επιτροπή Μεταφορών και ξέρω πόσο σημαντική είναι η αεροπορία όσον αφορά τον ανταγωνισμό, τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό. Το Συμβούλιο όμως επίσης πρέπει να δείξει καλή θέληση για να στηρίξει την αεροπορία. Κύριε Επίτροπε, σίγουρα γνωρίζετε ότι οι εξελίξεις στην αεροπορία επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Εσείς είπατε ότι χάνουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο επειδή δεν έχουμε πετύχει τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό όσο και η ασφάλεια των επιβατών. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξετε συγκεκριμένα μέτρα για τους ε, επιβάτες και την αεροπορία γενικότερα. Συμφωνώ λοιπόν με την στρατηγική σαν μια προσπάθεια να αποφύγουμε τα εμπόδια, αλλά θα ήθελα να δω στην πράξη πώ θα εφαρμοστεί. Θα υπερψηφίσω την έκθεση αυτή πάντω και ελπίζω όλε οι απόψει που ακούστηκαν εδώ σήμερα θα ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η νέα στρατηγική για τι αερομεταφορέ πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση τη βιομηχανία και του τουρισμού. Αυτό σημαίνει κυρίω μέτρα κατά των μονοπωλιακών καταστάσεων όπως αποτελεί η περίπτωση της fraport στην οποία παραχωρήθηκαν αντί πινακίου φακής δεκατέσσερα περιφερειακά αεροδρόμια στην ελλάδα και μάλιστα παραχωρήθηκαν με πρίκα μια και στα αεροδρόμια θεσσαλονίκης χανίων και σκοπέλου εκτελούνται έργα εσπα ύψους 520 εκατομμυρίων ευρώ γεγονός που απαγορεύεται από τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής ένωσης. επισημαίνεται ότι η fraport εκμεταλλεύεται το αεροδρόμιο της φραγκφούρτης και αεροδρόμια στα βαλκάνια δεδομένου ότι μέτοχος της fraport είναι η lufthansa καθίσταται σαφές ότι η fraport έχει πλέον μονοπωλιακή θέση στην ελληνική αγορά μετατρέποντας την ελλάδα σε γερμανικό τουριστικό προτεκτοράτο. πρόκειται για μια απεικιοκρατικού τύπου παραχώρηση ελληνικής δημόσιας περιουσίας σε γερμανική κρατική επιχείρηση στο πλαίσιο των μνημονιακών επιταγών. πρόκειται για παραχώρηση η οποία διαλύει τις εργασιακές σχέσεις και θέτει κρατικές υπηρεσίες στην υπηρεσία της fraport όπως δηλαδή συμβαίνει με την Πύρος Βεστική και το ΕΚΑΒΟ. υποστηρίζω κύριε πρόεδρε την τροπολογία για την κατάργηση της παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στη fraport. σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο κύριος Πιμέντα Λόπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Η στρατηγική αυτή είναι γεγονός ε, ότι δεν μας ικανοποιεί. Εμείς την καταγγέλουμε. Στόχο έχει ένα μονοπόλιο ε, και απώλεια εθνικής κυριαρχίας σε ένα σημαντικό στρατηγικό τομέα για την ανάπτυξη των κρατών μελών. Επίσης εντατικοποιεί την εκμετάλλευση των εργαζομένων που έτσι κι αλλιώς είναι στην επισφάλεια και χάνουν τους μισθούς τους. Ε, όλο και περισσότερο έχουν άτυπες λεγόμενες μορφές συμβάσεων ε, και οι μεγάλες εταιρείες αυτό ε, αποσκοπούν. Εμείς μιλάμε για να θεωρήσεις οδηγιών, για ε, να εθνικοποιείται η ζημία και να ιδιωτικοποιείται το κέρδος. Μόνο αυτό ενδιαφέρει τις μεγάλες εταιρείες, μεγιστοποίηση του κέρδους. Επίσης μας μιλούν για τον αντίκτυπο της απελευθέρωσης στη σχέση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Αλλά δεν προτείνουν απαντήσεις. Η μόνη απάντηση είναι άκρατη απελευθέρωση. Δικασία του Κατστιάη. Α, συγγνώμη. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Καπούτο, με τον οποίο ολοκληρώνουμε και τη διαδικασία του Κατστιάη. Κύριε Καπούτο, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, οι αερομεταφορές είναι ο κροκονίος λίθος για την κινητικότητα και έτσι υλοποιείται η ελευθερία διακίνησης όπως προβλέπει η συνθήκη. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς τα πρότυπα θα παραμείνουν υψηλά όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια και στην πτήση και στις υπηρεσίες υδάφους υπέρ των επιβατών και επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις ε, ψηφιακές τεχνολογίες. Έχουμε τον ε, ε, ενιαίο χώρο και θα πρέπει να αποφύγουμε τις αποκλήσεις από πλευράς κρατών μελών, να μην έχουμε τέλη και φόρους που ταλαιπωρούν τους πολίτες, αυξάνεται το κόστος, αλλά έχουμε τώρα και αύξηση του χρόνου πτήσεων και περισσότερη βλάβη στο περιβάλλον. Άρα χρειάζεται εξορθολογισμός. Ε, θα πρέπει αυτό να το κάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συνεχίσει να είναι η, ασφάλεια και η προσβασιμότητα η προτεραιότητα. Το λόγο έχει εξ ονόματος της Επιτροπής η Επίτροπος κυρία Μπούλτς. President. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, πολλά ζητήματα, πολλές ερωτήσεις. Όμως πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ του συζητητέ, τον κύριο Τάλιτσκα και τον κύριο Κρίστενσεν, για την τόσο πλήρη εκθεσή του. Και σα ευχαριστώ και για αυτή την τόσο καρποφόρα συζήτηση που είχαμε μαζί. Θα ήθελα να απαντήσω σε όλου σα, αλλά περιορίζει ο χρόνο, οπότε θα επικεντρωθώ σε κάποια ζητήματα και ελπίζω να μα δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε διμερό αργότερα για όλα τα ζητήματα που θίξατε. Πρώτα απ' όλα για τα βιοκαύσιμα. Στη στατηγική μας για χαμηλές εκπομπές Είμαστε σαφείς για το πόσο μεγάλη σημασία έχουν ενελεκτικές ενέργειες για τις μεταφορές. Για την αεροπορία τα βιοκαύσιμα είναι μια εναλλακτική που στηρίζουμε πλήρως. Όσον αφορά την πολυτροπικότητα και την ποιότητα του αέρος. Η πολυτροπικότητα σίγουρα είναι κάτι που έχει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ε, τοπικά. Οπότε θέλουμε να είναι πολυτροπικές οι λεωφόροι της αεροναυτιλίας. Θέλουμε επίσης να αναπτύξουμε συστήματα δημόσιων μεταφορών και υπέρ του περιβάλλοντος, αλλά και για να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός. Συνεχίζουμε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα για τα περιφερικά αεροδρόμια. Η θετικά ιδιαίτερα είναι όσον αφορά την τοπική οικονομία. Τα πρόσφατα χρόνια τα περιφερειακά αεροδρόμια ε, πηγαίνουν προς εμπορικούς στόχους και έχουν ανταγωνισμό μεταξύ τους για να προσελκύσουν κυκλοφορία. Σε αυτό το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρχει στρέβλος του ανταγωνισμού. Οπότε θέλω να αναφέρω εδώ τους κανόνες ε, δημόσιων ενισχύσεων που δεν πρέπει να πλήττουν τον ανταγωνισμό ούτε μεταξύ περιφερειακών αεροδρομίων. Οι μας γραμμές λένε πιο συγκεκριμένα κάτω από ποιε συνθήκες μπορεί να δικαιολογούνται τέτοιες κρατικές ενισχύσεις. Τώρα, για τα προγράμματά μας. Η Επιτροπή ξέρει ότι ένας τουλάχιστον διεθνής ε, εταίρος έχει συμμορφωθεί με το screening, δηλαδή με τους προελέγχους για τους επιβάτες, για τα στοιχεία των επιβατών έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος. Το θέμα αυτό του προλέγχου θα πρέπει να το κοιτάξουμε παρετέρω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης έχει σημειώσει ότι το αμερικανικό πρόγραμμα έχει σαν αποτέλεσμα να επιταχύνεται η διαδικασία προκειμένου να αφηχθεί κάποιος στις Ηνωμένε Πολιτείες. Έχουν έρθει σε επαφή με τις Αμερικανικές Αρχές για να δούμε αν μπορούμε και εμείς να εφαρμόσουμε ένα αντίστοιχο σύστημα. Να δούμε τι διαφορετικές αλλαγές θα πρέπει να γίνουν έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αυτός ο προέλεγχος λοιπόν είναι ένα θέμα που θα εξετάσουμε παρετέρω. Τώρα για το pay to fly. Όντω υπάρχουν τέτοια μοντέλα που αναπτύσσονται όσον αφορά το πλήρωμα. Να πληρώνει δηλαδή για να πετάξει. Είναι αρνητικέ οι επιπτώσει. Η Επιτροπή και, το, και η ΕΑΣΑ εξετάζουν αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι έχω εξαλείψει το χρόνο μου, οπότε για τα υπόλοιπα ζητήματα ευχαρίστω να τα ζητήσουμε διμερός. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την προσοχή σα και χαίρομαι πολύ που συμφωνούμε ότι θέλουμε να κάνουμε την αεροπορία μας μια ιστορία επιτυχή. Κυρία Επίτροπε, το λόγο έχει ο εισηγητής ο κύριος Τέλιτσκα για δύο λεπτά. Uh, by... Σας ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τους συναδελφούς Κλούν, Φώστερ, όλους με όσους ε, συνεργάστηκα. Ήταν ε, η συμβολή σας πολύ σημαντική. Κατά δεύτερο λόγο, να το πω για τις παρατηρήσεις κυρία Κονέτσνα. Είπατε ότι είναι σημαντικό το ότι τονίσαμε τα κοινωνικά θέματα, αλλά θυμηθείτε τι συζητήσαμε δεν είχατε μπορέσει να έρθετε σε καμία τη αντίστοιχη μα, Μα θα γνωρίζετε να ερχόσασταν ότι τα συζητήσαμε αυτά και τα συζητήσαμε ευθύ εξ αρχή. Και το πρόβλημά μου είναι ότι είχαμε τη γνωμοδέτηση τη Επιτροπή Απασχόληση που ήταν πάρα πολύ μακροσκελής. Οπότε ήταν δύσκολο όλα αυτά να τα καλύψουμε. Χρειάζεται κάποια πειθαρχία. Οπότε προσπαθήσαμε να τα συνοψίζουμε τους συναδέλφους. Οπότε πάντα είχαμε τα κοινωνικά θέματα στο επίκεντρο. Οι για τις στρατηγικές. Είπαμε να έχουμε μια στρατηγική, είναι πολύ σημαντική, αλλά και εκεί πρέπει να γίνουν κάποιες περικοπές, λάβαμε υπόψη ε, ό,τι χρειαζόταν, αλλά αν ήταν κάτι πολύ μακροσκελές, κανείς δεν θα τα διαβάσει. Οπότε και εγώ προσπάθησα να αναφέρω όλα τα μέσα, τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Αν κοιτάξτε τι γίνεται με τον δείκτη συνδεσιμότητας. Να, πώς μπορούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Κυρίε και κύριοι, έχω ένα όνειρο. Να ξυπνήσω μια μέρα, ένα πρωί και να αποφασίσω με την οικογένειά μου να πετάξω, να ταξιδέψω κάπου. Αλλά θέλω να υπάρχει αυτό το ολοκληρωμένο ενιαίο εισιτήριο που να με πάει από την Πράγα κάπου αλλού και μετά να πάρω το τρένο για να πάω στο χωριό μας ή κάπου αλλού σε ένα άλλο χωριό αυτό να είναι εύκολο να γίνει, να μην υπάρχουν όλες αυτές οι ταλαιπωρίες της ασφάλειας των προελέγχων, να μπορέσω να έχω μια πτήση, είτε είναι διεθνής, είτε είναι ευρωπαϊκή, να μην υπάρχει θόρυβος, να είναι το πλήρωμα ξεκούραστο, να μην γίνονται βλαπτικές εκπομπές, να μην υπάρχουν ανομαλίες με την κυκλοφορία των αεροδρομίων. Οπότε και αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι άλλο ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Είμαι σίγουρος ότι με τη δραστήρια ε, επιτροπή μας θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα.